η ουσία ουσιαστικά όπως προέκυψε τελικά ήταν ε, η ανάγκη στενή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ όλων των οργανισμών και μεταξύ όλων των κρατών μελών. Αυτή ήταν η ουσία που προέκυψε από αυτή την πρώτη έκθεση, ότι αυτή η συνεργασία είναι αναγκαία. Αν δεν υπάρχει αυτή η συνεργασία, τότε ό,τι μέτρα και να πάρουμε δεν έχουν νόημα ό,τι μέτρα να πάρουμε για οποιοδήποτε ε, κλάδο δεν χρησιμεύουν σε τίποτα αν δεν υπάρχει αυτή η συνεργασία μεταξύ όλων των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Ε, απομένουν ακόμα πολλά να γίνουν. Αυτό είναι ένα πόρισμα από τη δική μου έκθεση, διότι όπως το ξέρετε εσείς ε, και όσοι διάβασαν την έκθεση γνωρίζουν επίσης ότι ναι, έχουν γίνει μεν πάρα πολλά, έχουν επιτευχθεί πολλά, έχουν ε, ληφθεί πολλά μέτρα και εφαρμοστεί και αυτό είναι θετικό. Και η αρχή ΟΛΑΦ έχει οργανωθεί και δομηθεί πάρα πολύ καλά, αλλά ο αριθμός των υποθέσεων έμεινε απαράλλακτος. Και το ύψος της απάτης έχει ε, μεγαλώσει, έχει φουσκώσει σε τεράστιο βαθμό. Για μένα αυτό αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα και μήνυμα σημάδι ότι κάτι δομικά δεν πάει καλά και ότι έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης. Αυτό το λέω ξεκάθαρα και στην έκθεσή μου, ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στου θεσμού τη. Πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την εμπιστοσύνη των πολιτών προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι κοινή επιθυμία όλων. Αλλά πώ θα γίνει αυτό, πώ θα βελτιωθεί η εμπιστοσύνη όταν διαρκώ ακούγονται ε, σκανδαλώδεις υποθέσεις διαφθοράς ή ε, απάτης όπως ακούμε τώρα σε διάφορες χώρες ε, Υποθέσει που εξετάζουμε και εδώ στην ΚΟΝΤ. Όταν εμφανίζονται διαρκώς τέτοιες υποθέσει ε, που γίνονται πρωτοσέλδες εφημερίδες, φυσικά ε, υποβαθμίζουν και αποδυναμώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να μην αναλύσω ένα-ένα τα διάφορα σημεία που υπάρχουν μέσα στην εκθεσή μου, μπορείτε να τα διαβάσετε. Δεν σας λέω κάτι νέο ή έκθεση αυτή βασίζεται στις παλιότερες εκθέσεις. Δεν είναι ότι επινοούμε τον τροχό από την αρχή. Ε, απλά έχουμε συμπληρώσει κάποια πράγματα όπως είναι φυσικό και χαίρομαι φυσικά ε, και θα χαρώ φυσικά αν θεωρήσετε ότι ήταν ενδιαφέρουσα η έκθεση και μου κάνετε ερωτήσεις. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή θα μπορέσει ε, να χρησιμεύσει σε κάτι, να μας δώσει μια κατεύθυνση ε, αναφερόμαστε και στις ε, επιτυχίες φυσικά της Όλαφ και ελπίζουμε να τη βοηθήσουμε με αυτή την εκθέση και όπως είπα θα χαρώ να ακούσω τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας ε, ε, να συμβάλλετε όπως μπορείτε στη συζήτηση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Κούς για την παρουσίαση του εγγράφου σας. Συνεχίζω εγώ τώρα διότι η κυρία Χόλμαερ χρειάστηκε να, να αποχωρήσει. Λοιπόν, σας ξαναευχαριστούμε κύριε Κούς και δίνουμε το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές. Παρακαλώ περιοριστείτε στα τρία λεπτά για να τηρήσουμε τους χρόνους της συνεδρίασής μας. Δίνω λοιπόν πρώτα απ' όλα το λόγο στον κύριο Λέναρς για το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω σε τρία λεπτά. Είναι μια σημαντική έκθεση αυτή η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί είναι πολύ σημαντικό τα χρήματα τα οποία δαπανώνται από κοινού να δαπανώνται με καλό τρόπο και να φτάνουν στον προορισμό τους, στον πραγματικό. Πράγματι αυτό είναι ο μόνος ο τρόπος να έχουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Άκουσα την καρικατούρα πούμε, που είπε ο εισηγητής ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι πολίτες εξαιτίας αυτού. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν και στην Ολλανδία μάλιστα ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το Ισχύει αυτό στην Ολλανδία αλλά και σε άλλε χώρε, πιστεύω. Οπότε να μην υπερβάλλουμε αυτέ τι εκθέσει, να μένουμε στα σημαντικά. Και το σημαντικό εδώ είναι ότι το 2018, όπω και παλιότερα, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται η δαπάνη βάσει παρατυπιών. Οι διάφορες συναντήσεις που θα έχουμε και σήμερα το απόγευμα και αύριο και μεθαύριο και στο Σεβούλιο ξανά για τον προϋπολογισμό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ε, λιγότερες παρατυπίες κατά 2,5 δισεκατομμύρια. Θα βοηθούσε πολύ. Τώρα κάποια πιο συγκεκριμένα σημεία. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Η κυρία Ριβεζή στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ πριν από δύο εβδομάδες διαμαρτύρονταν για το γεγονός ότι οι χώρες μέλη δεν δίνουν, δεν βοηθούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν δίνουν δηλαδή εισαγγελίε προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι δυνατόν το πρωί να ασχολούνται με ευρωπαϊκά ζητήματα και το απόγευμα να ασχολούνται με εθνικά. Αυτό δεν θα είναι αποτελεσματικό. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χρειάζεται στήριξη από τις χώρες μέλη. Όσον αφορά τώρα την στρατηγική της Επιτροπής κατά των παρατυπιών, 12 μόνο χώρες μέλη έχουν υιοθετήσει την νέα στρατηγική που έπρεπε να ισχύει από τις 6 Ιουλίου του 2019. Πρέπει να βρούμε τρόπους να ενθαρρύνουμε και να πιέσουμε περισσότερες χώρες να συμμετέχουν και αυτές. Και λίγες είναι οι χώρες που έχουν εθνικές στρατηγικές αντιμετώπισης των απατών. Πρέπει να ψάξουμε και να βρούμε γιατί αργεί η υλοποίηση και γιατί δεν υπάρχουν εθνικές στρατηγικές καταπολέμησης της απάτης. Είναι βέβαια γενικότερο το θέμα του προπολογισμού, αλλά ε, το θέμα του Ταμείου επενδύσεων και επίσης και αυτό με απασχολεί. Τίποτα συγκεκριμένο δεν αναφέρεται. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις περιπτώσεις διαφθοράς, ας πούμε στη Γεωργία, στην Τσεχική Δημοκρατία. Καλό θα ήταν να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το naming and shaming, δηλαδή να κατονομάζουμε χώρες. Βλέπω ότι τέλειωσε ο χρόνος μου. Κάτι τελευταίο παρακαλώ. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά το βασικό πρόβλημα με τις εκθέσεις αυτές είναι ότι δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Και μετράμε τις παρατυπίες και τις απάτες έχοντας ελάχιστα ε, στοιχεία. Θα έπρεπε λοιπόν να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε διαφορετικά τα πράγματα και να δούμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την μεθοδολογία μας, ώστε ό,τι εντοπίζουμε να αντικατοπτρίζει το πραγματικό πρόβλημα, κάτι το οποίο δεν είναι βέβαιο τώρα. Ευχαριστώ για το χρόνο που μου διαθέσατε και εννοείται πριν υποβάλουμε τροπολογίες την επόμενη εβδομάδα θα ξανακοιτάξουμε το κείμενο. Ευχαριστούμε κύριε Λέναρς για τις παρατηρήσεις σας. Δίνουμε τώρα το λόγο στην κυρία Κρέτσου των Σοσιαλδημοκρατών. Σκιώδης επίσης η για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι η τριγωστή έκθεση που έχουμε για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια πολύ σημαντική έκθεση και αρκετά πλήρης και αναφέρεται στα έσοδα, στις δαπάνες και στην κατάσταση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. και τη διαχείριση που γίνεται σε αυτόν. Θέλω να προσθέσω στην έκθεση που έχουμε μπροστά μας, το σχέδιο έκθεσης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συντάσσουμε εμείς, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη γνώμη μου, δεν προστατεύει τελικά τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δούμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν πρόκειται για πάρα πολλά χρήματα τα οποία χάνονται από απάτες. Πρόκειται για ένα μικρό ποσό. όμως η έκθεση επικεντρώνεται υπερβολικά στα αρνητικά στοιχεία. Υπογραμμίζει τη λύπη στην νομοθεσία και με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι κάνει πιο έντονο το αίσθημα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήδη υπάρχει σε κάποιους πολίτες. Ήμουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ξέρω πολύ καλά ε, ότι γίνονται τεράστιες προσπάθειες για την καταπολέμηση της ε, απάτης. Το 0,5% απάτης δεν είναι κάτι που μπορεί κανείς να περιγράψει ως ε, τεράστια απάτη. Και εν πάση περιπτώσει τα χρήματα αυτά καλύπτονται από τις χώρες μέλη στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Έχουμε 4% σφάλματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς όμως οικονομικές επιπτώσεις. Υπογραμμίζω λοιπόν ότι ένα από τα κύρια συμπεράσματα ε, της έκθεσης 2018 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και που υπάρχει και στην ιστοσελίδα της Όλαφ είναι ότι πέρυσι είχαμε πρόοδο ώστε να δαπανώνται όλα τα ευρώ από τον κοινοτικό προπολογισμό καλά. Και υπάρχει ένα ισχυρό σύστημα προστασία του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Υπογραμμίζει επίση η έκθεση αυτή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλλον μιλάω για την έκθεση τη Όλαφ τώρα, που λέει ότι η Επιτροπή έχει οθετήσει μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης, για παράδειγμα και νέους απλοποιημένους κανόνες για τις δαπάνες από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και βελτιώνεται ο εντοπισμός, η ανείχνευση και η ανάκτηση κονδυλίων όταν υπάρχουν ε, απάτες. Και έτσι μειώνονται τα ποσά που χάνονται. Πρέπει να ενισχυθεί το σύστημα ακόμα περισσότερο και διαδικασίες, κυρίως όσον αφορά τον εντοπισμό και την ανείχνευση. Πάντως εμείς δεν βλέπουμε τίποτα τέτοιο στην έκθεση την οποία συντάσσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρόλο που ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόοδος αυτή. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να εντοπίσουμε πού βρίσκονται τα πραγματικά προβλήματα και να βρούμε λύση για να τα ξεπεράσουμε. Μην υπογραμμίζουμε μόνο τις αρνητικές πτυχές, χωρίς να κοιτάμε τη συνολική εικόνα της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια βελτιώνουν τα τελευταία χρόνια την ζωή των ανθρώπων σε 190 περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παντού βλέπετε νοσοκομεία, αυτοκινητόδρομους, παιδικούς σταθμούς, ε, ερευνητικά κέντρα, ένα σωρό προγράμματα. Ξέρετε, στην Ιταλία είχαμε και, και στην Πορτογαλία δείξαμε την αλλαγή μας απέναντι σε φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές κτλ. Και εκατομμύρια νέες θέσεις απασχόλησης δημιουργούνται με ευρωπαϊκή συνεισφορά. Γι' αυτό και εγώ είμαι έτοιμη να συντάξω ένα εναλλακτικό κείμενο για την Ολομέλεια. Και θέλω να καλέσω τους σκιώδες εισηγητές και ελπίζω και τον ίδιο τον εισηγητή να θέλει να συμμετάσχει σε μια συνάντηση ώστε να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς. Γιατί νομίζω ότι με αυτή τη λαϊκίστικη προσέγγιση παίζουμε με το μέλλον των παιδιών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Κρέτσου. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Ραμόνο Στρογγάριο του Ρινιού. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο παρακαλώ, περιοριστείτε, ε, κυρία Βουλευτή, παρακαλώ περιοριστείτε στα τρία λεπτά. Ευχαριστώ, θα μιλήσω ρουμανικά. Κύριε Πρόεδρε, θα περάσω αμέσως στο θέμα. Δυστυχώς, η ομάδα μας και το ραμά μας για την καταπολέμηση της απάτης δεν αναφέρεται παρκώς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το τι πιστεύει ο κόσμος. Αυτά απομακρύνονται πολύ από αυτά τα οποία λέει η έκθεση. Στην έκθεση γίνεται λόγος για 150 εκατομμύρια σε απάτες. Κάποιοι λένε ότι αυτά μπορούν να φτάσουν σε 900 εκατομμύρια στην πραγματικότητα. Το άρθρο 310 της συνθήκης μας δίνει την νομική δυνατότητα να καταπολεμήσουμε την απάτη και κάθε άλλη δραστηριότητα η οποία επηρεάζει πλήττει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Υπάρχουν δηλαδή οι αρμοδιότητες για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων. Ας, τα, ας τις αξιοποιήσουμε. Τα νούμερα αυτά δείχνουν ότι η διαστάση που έχει πάρει η απάτη κατά του ευρωπαϊκού προπολισμού έχει σταθεροποιηθεί, αλλά αν δούμε την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για το 2019, εκεί το ελεγκτικό συνέδριο έφτασε την προσοχή μας στα λίμματα του μηχανισμού ελέγχου για τον εντοπισμό της απάτης και από τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι μια σημαντική δυναμία. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την απάτη, ένα φαινόμενο σαν την απάτη, αν δεν έχουμε αίσθηση των πραγματικών διαστάσεων της απάτης, αν δεν κατανοήσουμε το φαινόμενο. Ακόμη και αν δεχθούμε ότι η απάτη μειώνεται τα τελευταία χρόνια, τα εν λόγω ποσά, τα καταδολιευόμενα ποσά, παραμένουν πολύ ψηλά, ειδικά στο Ταμείο Συνοχής. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να δραστηριοποιηθεί φέτος. Και χρειαζόμαστε και άλλες στοχευμένε πρωτοβουλίες για να ελοπίσουμε αυτήν τη δέσμευσή μας, την καταπολέμηση της απάτης. Και χρειαζόμαστε φυσικά και επαρκείς πόρους για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως είπα, η οποία θα δρομολογήσει τις σχετικές έρευνες. Αυτά χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης εκδίδει μια ετήσια έκθεση για την διαφθορά, άλλο ένα εργαλείο. Και με την ευκαιρία θέλω να καλέσω την Προεδρία του Συμβουλίου να μην δεχθεί στο πλαίσιο της σύντησης για τον προπολισμό συμβεσμούς όσον αφορά τον μηχανισμό που προτείνει η Κομισιόν για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων. Χωρίς αυτό δηλαδή να συνδέεται με το κράτος δικαίου. Σε κάθε περίπτωση για μας είναι μη διαπραγματεύσιμο το θέμα το θέμα τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων και όσον αφορά τη σύνδεση διαφθορά και προστασία οικονομικών συμφερόντων, κάτι πρέπει να κάνει η Κομισιόν, κάτι περισσότερο. Μόνο 11 από τα 27 κράτη-μέλη έχουν μια στρατηγική κατά τη απάτη και 12 μόνο μετέφεραν ικανοποιητικά τη σχετική οδηγία που αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτέ οι διαδικασίε πρέπει να επιταχυνθούν και όχι το αντίθετο, και να κινηθούν και διαδικασίε κατά των κρατών μελών που δεν, την, δεν τηρούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το ποσοστά λοιπόν εντοπισμού της απάτης είναι χαμηλά, ακόμη και σήμερα. Η Κομισιόν κάτι παραπάνω πρέπει να κάνει και χρειάζεται ε, γενικότερα ούτως ή άλλως μια πιο συντονισμένη προσπάθεια. Αυτά. Ε, κατά τα άλλα, συμφωνώ με τους ε, προλελήσαντες. Προτείνω, μάλιστα, να παρατείνουμε κατά μία τουλάχιστον εβδομάδα την προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Εγώ θα πρότεινα μάλιστα ένα εναλλακτικό ψήφισμα, ε, αν δούμε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Ευχαριστούμε πολύ. Δίνω το λόγο τώρα στον σκιώδη των Πρασίνων, τον κύριο Πέξ, παρακαλώ. Τρία λεπτά. Uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Κούς για μια ολοκληρωμένη έκθεση η οποία αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Θα λέγαω ότι χρειαζόμαστε κάποιες επιπλέον τροπολογίες. Συνεφώς υποστηρίζω την πρόταση της συναδέλφου να μεταθέσουμε την προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών κατά τουλάχιστον μία εβδομάδα. Θα ήθελα να θίξω τρία θέματα. Το ένα αφορά τις τροπολογίες, το άλλο αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θυμάστε τις απαλλαγές χθες. Με την ευκαιρία θέλω να τονίσω τη σημασία της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την αντιμετώπιση της απάτης και του διασυνοριακού εγκλήματος. Δυστυχώς πρέπει να επικρίνω για άλλη μια φορά την λυπή χρηματοδότηση και λυπή στελέχωση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Νομίζω ότι η Κομισιόν υποεκτίμησε με μεγάλη διαφορά τις πραγματικές ανάγκες. Από ό,τι φαίνεται η εισαγγελία θα έχει περίπου 3.000 επιπλέον υποθέσεις κάθε χρόνο. Η κυρία Ριβάση, μάλιστα πριν από μερικές εβδομάδες, είπε ότι κάποια κρατημέλη ε, έχουν σκοπό να διορίσουν εισαγγελής μερικής απασχόλησης. Αυτό είναι απολύτως ανεπαρκές και δεν διασφαλίζει για την ε, ανεξαρτησία τους. Να υπενθυμίσω σε όλους ότι πέντε χώρες ακόμη δεν έχουν, ε, ας πούμε η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σουηδία για παράδειγμα, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρέπει να το κάνουν αυτό, να συνταχθούν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το συντομότερο δυνατόν. Το δεύτερο πολύ σημαντικό που πρέπει να συζητήσουμε είναι η κατάχρηση στα γεωργικά ταμεία το φαινόμενο είναι συστημικό πρόβλημα. Η απάτη στον γεωργικό τομέα αυξήθηκε σε σχέση με πέρσι 10%. Πρόκειται για εκατομμύρια. Η Κομισιόν πρέπει να προτείνει τροποποίηση των, των κανόνων της ε, ΚΑΠ για να ενισχυθούν τα μέτρα ελέγχου για την πρόληψη της απάτης και τα κτηματολόγια να γίνουν πιο διαφανή. Όπως έγραψαν και οι New York Times, το κράτος δικαίου στην Ευρώπη σήμερα δεν έχει κανένα αποτέλεσμα στον γεωργικό τομέα, διότι οι ολιγάρχες ε, σφετερίζονται τη γη των μικρών παραγωγών, των μικρών αγροτών για να κερδίσουν στην Τσεχία, στην Ουγγαρία, στην, στην Πολωνία. Απογοητεύτηκα επίσης γιατί διάβασα ότι μόνο 12 κράτη-μέλη εφαρμόζουν πλήρω τη νέα οδηγία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποτίθεται ότι η προθεσμία ήταν πέρσι τον Ιούλιο και μόνο 11 κράτη-μέλη έχουν θεσπίσει, έχουν δημιουργήσει μια εθνική στρατηγική κατά τη απάτη. Καλό λοιπόν τα κράτη-μέλη να δράσουν το συντομότερο δυνατόν, συμπεριλαμβανομένη και τη δική μου χώρα, τη ε, Τσεχία. Θα καταθέσουμε λοιπόν τροπολογίες, όπως ε, προείπα, και θα ήθελα να έχουμε την ευκαιρία να τις ε, κρατήσουμε εγκαίρως. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πέξ. Τώρα είχαμε προβλέψει τους άλλους δύο σκιώδεις για το ECR και την ΚΟΕ, αλλά δεν βρίσκονται εδώ. Αφού μας μένει λοιπόν λίγος χρόνος, θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, αν υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να παρέμβει για να σχολιάσει, να ρωτήσει κάτι. Δεν υπάρχουν ερωτήσει. Ωραία. Δίνω λοιπόν το λόγο στην κυρία Μαργαρέτα Χοφμάν, Διευθύντρια Πολιτικής του Όλαφ, για να ακούσουμε τα δικά της ε, σχόλια. Σας, ε, θα σας παρακαλούσα να περιοριστείτε στα πέντε λεπτά. Έχετε το λόγο κυρία Χόφμαν. Yeah, thank you very much, ε, Mrs. Chair. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή για την έκθεσή του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα φαινοείται ε, πάντα θέλουμε να σας στηρίξουμε, να βοηθήσουμε και να εξηγήσουμε διάφορα ζητήματα, γιατί δεν είναι μόνο πολιτικό το θέμα, μερικές φορές είναι και τεχνικό. Επίσης, ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις των ε, σχεδόν εισηγητών με τους οποίους επίσης προσβλέπουμε συνεργασία, να δούμε τις τροπολογίες τους κλπ. Λοιπόν, το σχέδιο αυτό έκθεσης αποτελεί ήδη μια καλή βάση, πιστεύουμε, για να προχωρήσει βέβαια παρετέρω. Ήδη η έκθεση αναφέρει μερικά σημαντικά ζητήματα. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω πρώτα κάποιες γενικές παρατηρήσεις και μετά θα απαντήσω και στα ζητήματα που έθεσαν οι ευρωβουλευτές. Πρώτα απ' όλα, έγιναν διάφορες παρατηρήσεις όσον αφορά τη συνεργασία των χωρών μελών σε διάφορα επίπεδα και για τον ρόλο που παίζουν οι χώρες μέλη. Η έκθεση αυτή, πάνω στην οποία ε, συντάσσεται η δικιά σας έκθεση, αναφέρεται και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο επίπεδο χωρών μελών πώς μπορεί να καταπολεμηθεί δηλαδή η απάτη ε, σε βάρος του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να καταδείξει ότι γίνονται από κοινού προσπάθειες, ότι ήδη δηλαδή υπάρχουν πολλά μέτρα που έχουν υιοθετήσει οι χώρες μέλη κατά το παρελθόν, τα τελευταία χρόνια. Το λέμε στην έκθεσή μας ότι οι προσπάθειες γίνονται από κοινού με τις χώρες μέλη. Η έκθεση λοιπόν είναι μια καλή έκθεση δείχνει την ε, βούληση καταπολέμησης της απάτης. Φυσικά όλοι γνωρίζετε ότι υπάρχουν προβλήματα και αυτά θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Η έκθεση λοιπόν σε αυτό ακριβώς συνεισφέρει. Τώρα για κάποια θέματα που θίξατε εσείς. Ας αρχίσω από κάτι που αναφέρθηκε πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την επάνδρωσή της με αρκετό προσωπικό, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει πλήρως από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, δηλαδή από τα τέλη αυτής της χρονιάς. Όλοι γνωρίζουμε, το ξέρετε ότι υπάρχουν περιορισμοί οικονομικοί, αλλά πιστεύουμε ότι τελικά θα βρεθεί μια καλή λύση που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αναλάβει τα καθήκοντά της συγχρόνως με την Όλαφ για να έχουμε σώματα ισχυρά που να καταπολεμούν την απάτη, τη διαφθορά και την εγκληματική συμπεριφορά στην Ευρώπη. Και αυτό με διοικητικά μέτρα ανάκτησης κονδυλίων αλλά και πρόληψης. Τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Ε, σύμφωνα με την ρύθμιση μπορεί να υπάρχει μια τέτοια περίπτωση εισαγγελή να ε, απασχολούνται με μερική απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποιες μικρές χώρες που μπορεί να μην έχουν πολλές περιπτώσεις και ίσως ε, να μην ε, χρειάζεται πολλή απασχόληση από τη δική τους την πλευρά, αλλά θα το δούμε αυτό. Όσον αφορά την οδηγία, ναι, οι χώρες μέλη πρέπει να επιταχύνουν την ε, ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο. Όπως έχει ήδη υποθεί, μένουν πολλά ακόμα να γίνουν. Συνεργαζόμαστε με τις χώρες ε, μέλη και η Γενική Διεύθυνση Justice, Δικαιοσύνης και εμείς ε, πηγαίνουμε και προσπαθούμε να πιέσουμε ώστε να μπορέσει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ξεκινήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Σίγουρα θα υπάρξουν και διαδικασίες επί παραβάση. Τώρα, όσον αφορά τις εθνικές στρατηγικές καταπολέμησης της απάτης. Για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό και για την Επιτροπή και για την Όλαφ. Δεν υπάρχει όμως δυστυχώς υποχρέωση νομική ώστε να έχουν τέτοια στρατηγική οι χώρες μέλη. Κάποιες βέβαια έχουν και υπάρχει και διάσκεψη που προβλέπεται ώστε να βοηθήσουμε τις χώρες μέλη να προχωρήσουν στην υιοθέτηση μιας τέτοιας στρατηγικής καταπολέμησης της απάτης. Έγιναν και άλλες σημαντικές παρατηρήσεις και επανέρχονται κάθε χρόνο για το επίπεδο της απάτης γιατί το θέμα των ε, παρατυπιών ε, βέβαια ε, έχει να κάνει με το τι εντοπίζουν οι χώρες μέλη και τι μας μεταφέρουν εμάς. Η συζήτηση γίνεται πάντα. Πάντως με την στρατηγική της Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης που υιοθετήθηκε τον Απρίλιο που μας πέρασε, κάνουμε σε βάθος ανάλυση και λαμβάνουμε υπόψη μας περισσότερα στοιχεία για να έχουμε μια πιο ρεαλιστική εικόνα των των παρατυπιών που εντοπίζονται στις χώρες μέλη. Να ξέρετε πάντως πώς θα ενισχύσουμε τη συλλογή δεδομένων αναχώρα. Ξέρω ότι ξεπέρασα το χρόνο μου, γι' αυτό θέλω να ελέγξω εδώ τι έχω αφήσει. Όχι, νομίζω ότι αυτά είναι τα κύρια σημεία που ήθελα να σας μεταφέρω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Χόφμαν για τις ε, σκέψεις σας και για τις αναλύσεις που μας κάνατε σε σχέση με τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Θα ήθελα να ζητήσω από τον εισηγητή, τον κύριο Κούς, ε, αν θέλει να παρέμβει, να μας πει κάποια τελικά σχόλια σε σχέση με τα όσα υπόθηκαν ήδη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε ξανά τη δυνατότητα να απαντήσω σε κάποια πράγματα. Πριν κλείσουμε ήθελα να πω ότι οποιασδήποτε δηλώσεις υπάρχουν ε, και ισχυρισμοί υπάρχουν μέσα στην εκθεσή μου βασίζονται σε πράγματα ε, που έχουν υποθεί από την Κομισιόν, από τις αρχές της Όλαφ. Δεν ε, επινόησα κάτι, ούτε προσπάθησα να συμπεριλάβω πολιτικές σκέψεις. όλα οι πληροφορίε είναι τεχνικές. Οπότε δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί ε, θα πρέπει να αντικατασταθεί η εκθέση από κάποια άλλη. Εντάξει, η Επιτροπή θα το αποφασίσει. Σε ένα πράγμα, πράγμα ήθελα να εστιαστώ το οποίο δεν αναφέρθηκε. Εκεί που διακρίνω εγώ κάποιο πρόβλημα είναι ότι η υποβολή εκθέσεων, η σύνταξη εκθέσεων σε όλα τα κράτη-μέλη υπάρχει ένα όριο των 15.000 ευρώ. Δηλαδή όλες οι υποθέσεις απάτης και τα προβλήματα που είναι κάτω των 10.000, συγγνώμη, όχι 15.000 ευρώ, δεν ε, ε, περιλαμβάνονται στην ανάγκη υποβολής έκθεσης. οπότε όταν έχουμε μικροποσά κάτω των 10.000, αυτά διαφεύγουν. Είναι άγνωστο, άγνωστο η περιοχή αυτή. Δεν ξέρουμε σε τι συνίστανται αυτές οι απάτες και αυτό είναι δομικό πρόβλημα Όταν ξέρει δηλαδή κανείς ότι κάτω από τα 10.000 ευρώ δεν πρόκειται να τον βρουν, ούτε υπάρχει υποχρέωση υποβολής έκθεσης, ε, τότε θα ξεφύγει και αυτό για μένα ένα πρόβλημα. Τέλος, θέλω να σας πω μια μικρή ιστορία, η οποία ίσως δείχνει ε, σε τι συνίσταται η όλη κατάσταση. Ουσιαστικά, πριν από 250 χρόνια, στη Γερμανία ζούσε ο παλιός Φρίτσοφ, ο ο Φρυδερίκο ο Μεγάλο, ο βασιλιά τη Προσία, ο οποίο είχε ένα στρατηγό, τον Γιώχιμ Φοντσίτεν, και αυτό ο στρατηγό ήταν πολύ γνωστό τότε, πολύ πλούσιο και πολύ διακριτικό και είχε όλε τι προσικέ ε, αρετέ, όπω λένε. Και ένα βράδυ ήρθε να τον επισκεφθεί κάποιο φίλο και αυτός βρισκόταν απασχολημένο στο γραφείο του όπου υποδέχθηκε και τον καλεσμένο και εκεί έκαιγε η λάμπα, η λάμπα λαδιού πάνω στο γραφείο του και του λέει λυπάμαι, χρειαζόμαι ακόμα 15 λεπτά, λίγο κάτι να τελειώσω, ε, να κάνω μια δουλειά και συνεχίζει να δουλεύει και όταν τελείωσε έσβησε τη λάμπα, έσβησε τη φλόγα και άναψε μια άλλη λάμπα και του λέει ο φίλος του «Μα τι κάνεις εκεί» και αυτός λέει Δεν μπορώ να καίω το λάδι του βασιλιά μου για τις ιδιωτικές μου υποθέσεις. Αυτή η στάση, αυτή η συμπεριφορά σήμερα πιστεύω λείπει μερικές φορές. Όταν έχουμε αυτή την έκθεση πύφη η οποία ε, πρέπει να ενισχύσει αυτή τη συνείδηση ότι δεν μπορούμε εμείς να πλουτίζουμε από χρήματα κοινά που υπάρχουν για όλου. Ε, δεν είτε είναι του βασιλιά μα, είτε τη κυβέρνησή μα, τη δημοκρατία. Δεν έχει σημασία. Εάν αυτό δεν επιτύχει ως νοοτροπία θα αποτύχουν όλα μας τα μέτρα. Απλά θα τρέχουμε εμεί διαρκώς πίσω από ανθρώπους και θα καταλήγουμε σε διάφορα πορίσματα και θα καταλήγουμε πάντα στο ίδιο. Και η επιθυμία μου είναι, είναι φυσικά ευσεβής πόθος ίσως και μια πίστη δική μου ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση δίνοντας και εμείς το παράδειγμα ως ευρωβουλευτές όσον αφορά αυτή τη συμπεριφορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κούς για τα συμπεράσματα αυτά και για αυτή την πολύ ωραία ιστορία που μας είπατε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους οι οποίοι προενέβησαν σε αυτή τη συζήτηση διότι πιστεύω ότι οι σκέψεις που ακούσαμε και τα σχόλια μαρτυρούν όχι μόνο τη σπουδαιότητα αυτού του θέματο, ε, την υπεράσπιση των οικονομικών συμφερόντων τη Ένωση και την καταπολέμηση τη απάτη, αλλά και τη δέσμευση που πρέπει να δείξει όλο το Κοινοβούλιο, ούτω ώστε τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και κατ' επέκταση των πολιτών μας να ε, προστατευτούν αποτελεσματικά. Για να δεχτούμε τώρα το αίτημα που ακούσαμε στη διάρκεια της συζήτησης, ε, αποφασίσαμε να αναβάλουμε την προθεσμία υποβολή τροπολογιών είχε προβλεφθεί για 25 Φεβρουαρίου του 2020 αναβάλλεται για την 3 Μαρτίου του 2020 στις 2 το μεσημέρι. Ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση. Κλείνουμε αυτό το θέμα και πάμε στο επόμενο στη συζήτηση που ακολουθεί. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο της ημερής σας διάταξης Σήμερα είναι ο έλεγχο τη ε, έκθεση ιδέα πρωτοβουλία για τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι η ετήσια έκθεση του 2018. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η ΕΤΕ παίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών μεταξύ, μέσω διαφόρων εντολών ε, διαχείρισης, εργαλείων και δημοσιονομικών μέσων. Και επίσης θα χρησιμεύσει ε, για την υλοποίηση του σχεδίου Juncker, του ε, Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Sí. Possiamo, chiedo scusa un attimo. <laughs> Λοιπόν, είμαι βέβαιη ότι η ΕΤΕ θα συνεχίσει να παίζει ρόλο κλειδί και στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο από το 2021 μέχρι το 2027. Συμφωνούμε όλοι ότι αυτός όλο ένα και αυξανόμενο ρόλο τη ΕΤΕ θα πρέπει να εξετάζεται τακτικά από την Επιτροπή μα, αλλά και από το ελεγκτικό συνέδριο. aggiustamento. Ε, ζητώ συγγνώμη, είχαμε μια μικρή τεχνική προσαρμογή. Ήθελα λοιπόν να δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Έκχαουτ, στον οποίο θα ήθελα να ζητήσω να περιορίσει την παρουσίασή του, αν είναι δυνατόν, στα 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ, έχετε το λόγο. Thank you very much, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω σε 10. Μιλούμε για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την ΕΤΕΠ. Έχουμε το σχέδιο έκθεσης για τις ε, δραστηριότητές της. Συνέταξα σχέδιο έκθεσης που ακολουθεί τη συνήθη συλλογιστική. Ξεκινώ λέγοντας ότι Μιλούμε για το 18. της επιδόσεις το 18. Είμαστε ήδη βέβαια στο 20. Οπότε, ξέρετε, δύσκολα κρατείται κανείς το 18 ως ισχυτής, γιατί έκτορα έχουν συμβεί διάφορα. Μπορεί να δείτε κάποια ευελιξία όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο αναφορά στην έκθεση, το καταλαβαίνετε καταλαβαίνει και η τράπεζα, αλλά συμβαίνουν πολλέ αλλαγέ αυτή τη στιγμή στην τράπεζα, σημαντικέ για μα, για το Κοινοβούλιο, για την Επιτροπή μα. Έχουμε λόγο εφόλη τη ύλη. Ό,τι πούμε ε, θα έχει επιπτώσει και στο μέλλον τη ΕΤΕΠ. Α δούμε. Ξεκινούμε με μια σχετικά στεγνή αξιολόγηση των επιδόσεων, τη γεωγραφική κατανομή των συμβάσεων, ποιες χώρες υποφελούνται κατά κύριο λόγο. Εδώ χρειάζεται περαιτέρω εμβάθυνση και η ΕΤΕΠ πρέπει να το κάνει αυτό. Να δούμε τις χώρες, το κατακεφαλήν εισόδημα, της, το χάσμα των επενδύσεων από χώρα σε χώρα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Ξέρουμε ότι δεν είναι όλες οι χώρες ίδιες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, κύριες προτεραιότητες επενδυτικής πολιτικής Είμαστε τώρα στο μέσο της συζήτησης της τράπεζας που θα γίνει η τράπεζα για το κλίμα. Αυτή είναι και η φιλοδοξία της ίδιας της τράπεζας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας. Τονίζει συνεχώς ότι αυτό είναι σημαντικό και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, να γίνει η τράπεζα, να γίνει η ΕΤΕΠ, ε, η Πράσινη Τράπεζα, μια τράπεζα για το κλίμα. Είναι προτεραιότητα και της ε, Κομισιόν και της Επιτροπής. Αυτό που έχει σημασία είναι το πώς θα υλοποιήσει αυτόν ή μάλλον αυτούς τους στόχους η ΕΤΕΠ. Στόχος είναι όλες οι χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες να συνάδουν με το Παρίσι, 50% των επενδύσεων να συνάδουν ή να διευκολύνουν την ε, αηφορία, με στόχο να κινητοποιήσουμε συνολικά μέχρι το 2030 ένα 3 εκατομμύριο ευρώ για το κλίμα, που είναι και η φιλοδοξία της Επιτροπής. Τώρα, πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο του υπολογισμού, τι σημαίνει κλίμα, τι σημαίνει περιβαλλοντική αηφορία κλπ. Η ΕΤΕΠ έχει κάνει αρκετή δουλειά επί του θέματος. Καλό είναι όμως να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Επίσης έχει σημασία να συμφωνήσουμε τι σημαίνει, τι όταν λέμε να συνάδουν όλα αυτά με το Παρίσι, με τη Συμφωνία των Παρισίων, γιατί και εκεί υπάρχει αρκετό νερό και υπάρχει και περιθώριο βελτίωσης. Κοιτάζω λίγο, ξέρετε, προς τα αριστερά μου, γιατί εκεί είναι οι άνθρωποι της, ε, της ΕΤΕΠ. Λοιπόν, ναι, όχι, εντάξει, έχει κι άλλους, είναι χιλιάδες, αλλά... <laughs> Σχολιάζω επίσης την πολιτική δανείων στον ενεργειακό μεταξύ άλλων τομέα. Τονίζω και αυτήν, αυτόν τον τομέα γιατί ε, σε λίγο θα έχουμε να συζητήσουμε και τον τομέα των μεταφορών. Στη συνέχεια στην έκθεση προχωρούμε με τη συνεργασία της ΕΤΕΠ με την EBRD και τις άλλες αναπτυξιακές τράπεζες, πώς μπορεί αυτή η συνεργασία να βελτιωθεί για τους σκοπούς της ε, καλύτερης απόδοσης. Μετά σχολιάζουμε την χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση εν ώψη και του σχεδίου Juncker. Υπάρχουν θέματα διακυβέρνηση, όπω καταλαβαίνετε, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωση και της ΕΤΕΠ. Και, και αυτό είναι σημαντικό, και τονίζω επίσης ότι από πολιτική απόψεως υπάρχει πίεση να πετύχουμε κάποια επίπεδα χρηματοδότησης χάρη σε ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, χάρη σε μόχλευση, όμως από την τραπεζική άποψη το θέμα είναι Πού πρέπει πραγματικά να επενδύσουμε, πού υπάρχει έλλειψη επενδύσεων. Αυτό ήταν και το σχέδιο Juncker. Το λέω αυτό γιατί σε μερικέ περιπτώσει ε, δώσαμε την εντύπωση απλώς, ότι πρέπει απλώ να πιάσουμε ένα νούμερο. Και ήταν αυτό σημαντικό για το σχέδιο Juncker, αλλά ήταν σαν είχαμε αφήσει απ' έξω την ΕΤΕΠ. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε τα χάσματα, να επενδύσουμε εκεί που υπάρχουν ελλείψεις και το λέω αυτό στο κείμενο της έκθεσης. Και συνεχίζουμε με την διακυβέρνηση και τη δομή της σχολιάζω το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εταιρική διακυβέρνηση της ΕΤΕΠ, το πλαίσιο ελέγχων. Λέμε εδώ ότι αν δει κανεί τη διαφοροποίηση των έργων και την ανώτερη διοίκηση της ΕΤΕΠ, ε, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Πρέπει να το δηλαδή αυτό σοβαρά υπόψη της ΕΤΕΠ. Είναι αυτό που είχαμε δει ότι όταν ε, με την πολιτική δανείων στον τομέα τη ενέργεια. Επίση, στον τομέα τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και, και εκεί έχουμε περιθώρια βελτίωση. ειδικά επειδή η ΕΤΕΠ βρίσκεται στο κέντρο του δημοσίου διαλόγου αυτόν τον καιρό. Πριν λίγο καιρό κανεί δεν ήξερε ότι καν υπήρχε η ΕΤΕΠ, αλλά αυτά ανήκουν πια στο παρελθόν και αυτό είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Τα αιτήματα όμω περί διαφάνεια και λογοδοσία είναι πολύ πιο έντονα από την κοινωνία και αυτό αφορά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί του λαού τη Ευρώπη. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη διαφάνεια εναντί και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εν συνεχεία, στην έκθεση, σχολιάζω συστάσεις της Όλαφ, καταπολέμηση της απάτης, αντιμετώπιση των περιστατικών απάτης, ε, και εκεί υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Και τέλος, στην έκθεση πάντα καλούμε την ΕΤΕΠ να συνεχίσει να δημοσιεύει στοιχεία βάσει των προηγουμένων συστάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί διατυπώνουμε συστάσεις εδώ και καιρό και μας ενημερώνει κάθε τόσο η, ΕΤΕΠ πώς και τι κάνει, πώς βελτιώνεται, πώς υλοποιεί τις συστάσεις αυτές. Και τέλος, τέλος, λέμε ότι θα στείλουμε την έκθεση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, αλλά θυμίζουμε ότι τα περισσότερα θα συζητηθούν μεταξύ Συμβουλίου και Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕΠ. Θέλουμε να προκαλέσουμε αυτήν την συζήτηση λοιπόν. Εξού και η καταληκτική παρατήρηση στην έκθεση. Αυτά λίγο πολύ. Αυτά είναι τα βασικά ή τα, κύρια σημεία, εν πάση περιπτώσει, της ε, έκθεσης. Οπότε περιμένω με πολύ ενδιαφέρον τα σχόλια των σκιωδών και των άλλων συναντέλφων και βεβαίω και μια πρώτη απάντηση από την ΕΤΕΠ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Έικχουτ. Δεν φτάσετε τα 10 λεπτά που είχαμε προβλέψει. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και για την παρουσίαση του σχεδίου εκθεσής σας που πραγματικά πραγματεύεται πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Θα ήθελα να ζητήσω από τους κοιόδες τώρα να παρέμβουν για το ΕΛΚΑ. δεν βρίσκεται εδώ ο κύριος Βίντσεκ ο κύριος Στεχόφσκι παρακαλώ για τρία λεπτά Ευχαριστώ, πολύ δεν είμαι σκιώδης συζητητής, αλλά άμα χρειάζεται κάποιον ε, ισχυρό εδώ πέρα για να αντιταθεί στην έκθεσή σας εντάξει μου έδωσε τις παρατηρήσεις της ε, η σκιώδηση εισηγήτριά μας. Τέλος πάντων, πλάκα κάνω με αυτά που λέω. Λοιπόν, θα ήθελε να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την εξαίρετη πρότασή του και έχει κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτη παρατήρηση. Θα ήθελε να τονίσει ότι τα κλιματικά ζητήματα δεν λύνονται χωρίς στήριξη από την βιομηχανία. Οι αλλαγές θα μπορέσουν να ελοπιθούν μόνο αν και η βιομηχανία συμμετέχει και να προτείνει καινοτόμε λύσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Δεύτερον, Το να φύγουμε από τον άθρακα και τα αστερά καύσιμα, αυτό σταδιακά μπορεί να γίνει μόνο. Γιατί υπάρχουν ήδη συμβάσεις που τρέχουν. Έπειτα, θέλει να ξέρετε ότι το ΕΛΚ πιστεύει πως πηγές όπως το φυσικό αέριο συνεχίζεται στο δρόμο προς την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Επίσης, η υποχρέωση δημοσιοποίησης της έκθεσης σε στερεά καύσιμα δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος της πρόσβασης σε χρηματοδότηση όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τη διαφάνεια, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει αναλάβει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα έπρεπε να υπάρχει μια καλή ισορροπία ανάμεσα στα μέτρα διαφάνειας από τη μία και από την άλλη μεριά την γραφειοκρατία που επιβάλλεται. Επίσης η κυρία Βίνσικ θα υποβάλει κάποιες τροπολογίες ακριβώς για αυτά τα θέματα και θέλει και πάλι να σας ευχαριστήσει για το έργο σας και για τη συνεργασία σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Στεχόφσκι. Δίνω το λόγο στους σοσιαλδημοκράτες, την κυρία Κρέτσου, παρακαλώ για τρία λεπτά. Thank you, ε, also... Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι η έκθεση αυτή για τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι η τράπεζα αυτή έχει εξελιχθεί στο χρηματοοικονομικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδια για την υλοποίηση όλο ένα και πιο ποικιλόμορφων εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών. Χαίρομαι που βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει παράσχει πάνω από 64,9 ε, δισεκατομμύρια ευρώ για ε, χρηματοδότηση με υπογραφή 854 έργων. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπάσα Εκχουτ, τον εισηγητή, για την έκθεση αυτή, που αποτελεί πολύ καλή συνέχιση της ε, περσινή έκθεσης. Ωστόσο, ως πρώην ε, Επίτροπος Περιφερειακών Θεμάτων παρατήρησα ότι στο πρώτο κομμάτι ξεχάστηκε η συνοχή παρότι πάνω από το 33% της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είχε περισσαφιερωθεί στην συνοχή. Οπότε εμείς ως σοσιαλδημοκράτες θα υποβάλουμε τις σχετικές τροπολογίες, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο ρόλο έχει παίξει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και πώ έχει αυξηθεί αυτό ο ρόλο στην πολιτική συνοχή στα τελευταία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει δώσει δάνεια για επενδυτικά προγράμματα σε λιγότερο ανεπτυγμένε περιοχέ, συχνά με χρηματοδότηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ούτω ώστε να προσελκύουμε και άλλου επενδυτέ. Φυσικά το πρασίνισμα τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επίση είναι θέμα ευρεία συζήτηση σήμερα. Αυτό τονίζεται φυσικά στην έκθεση, αλλά όπως είπα δεν μπορούμε να ξεχνάμε τις προτεραιότητες της ε, τράπεζας όπως, ε, της τράπεζας όπως θεσπίζονται στη συνθήκη. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των αναπτυγ... λιγότερων αναπτυγμένων περιοχών. Σύμφωνα με το άρθρο 309 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να υποστηρίζει και έργα για την ανάπτυξη λιγότερων αναπτυγμένων περιοχών. Όπως είπα λοιπόν, πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να μην αφήσουμε καμιά περιοχή να μείνει πίσω και να καταβάλουμε περαιτέρω προσπάθειες για τη μείωση των ανισοτήτων. Φυσικά οι κλιματικοί στόχοι είναι πολύ σημαντικοί για την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων πρέπει να ε, ευθυγραμμίζονται και με τη Συμφωνία του Παρισιού αλλά δεν μπορούμε να παραδεχτούμε ότι οι κλιματικοί στόχοι εντείνουν τις διαφορές μεταξύ περιφερειών και χωρών. Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ για το πώς θα το διατυπώσουμε αυτό. Πρέπει να συνδυασούμε σωστά τις παλιές με τις νέες προτεραιότητες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κρέτσου. Δίνω το λόγο στον κύριο Κριστιαν Κινέα από το Ρήνιου. Έχετε τρία λεπτά. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, κύριε Σιγητά, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Τέσσερα θέματα θέλω να καλύψω. <clears throat> Πρώτον, πιστεύω ότι είναι καλό στην έκθεση αυτή το ότι θέλει η τράπεζα να επικεντρωθεί σε μικρά και μεσαία προγράμματα και σε πρωτοβουλίες των πολιτών. Είναι κάτι που μας βρίσκει σύμφωνος. Δεύτερον, το κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται στο μηχανισμό για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς. Η τράπεζα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη συνεργασία και με την Όλαφ και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι καλό και αυτό το κεφάλαιο. Τρίτον, όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή. Εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν ε, διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ έχω υπολογίσει ότι το 2018, αν δούμε γεωγραφικά τις διάφορες συμβάσεις, πέντε υποφελούνται κυρίως από τις χώρες μέλη. Με 52, ενώ το 2017 είχαμε 54. Η εξέλιξη δηλαδή δεν είναι σημαντική και θα ήθελα αυτό να τονίσετε περισσότερο. Δηλαδή το ότι υπάρχει μια γεωγραφική ανισορροπία η οποία παραμένει. Το σχέδιο έκθεσης επίσης επιμένει για το ότι πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τους κλιματικούς στόχους η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και επιμένει πολύ από αυτού. Εγώ όμως πιστεύω ότι εδώ αναφέρονται κάποιες υπερβολές. Για παράδειγμα, στην παράγραφο 20 λέει ότι καταδικάζει το γεγονός ότι το 2018 ενέκρινε κάποια σχέδια η τράπεζα Αζερβαϊτζάν, Ανατόλια κτλ. Όπως επίσης και αυτό που συνδέει την Ελλάδα με την Ιταλία μέσω της Αλβανίας και της Αδριατικής θάλασσας. Είναι παράγραφος 21. Όντω πρόκειται για σχέδια κοινού ενδιαφέροντος. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μάλιστα, πριν από δύο εβδομάδες τα είχε συμπεριλάβει στο τρέχοντα κατάλογα. Είναι υπερβολή δηλαδή να λέμε ότι λυπούμαστε για το γεγονό ότι η τράπεζα χρηματοδοτεί αυτά. Τώρα επειδή είμαι και αντιπρόεδρο στην Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων και είχαμε και εκεί συζήτηση για το κατά πόσο οι χώρε μέλη πρέπει ή όχι να χρηματοδοτούν ε, από το Ταμείο Συνοχής ε, προγράμματα που έχουν να κάνουν με το φυσικό αέριο. Συμφωνώ ότι μεταβατικά μπορεί να γίνεται αυτό, σαν μια μεταβατική δηλαδή πηγή ενέργειας, χωρίς να λέμε ότι αυτό αντιβαίνει στους στόχους για καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Θα υποβάλω λοιπόν κάποιες τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε κύριε Γκινέα. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Τζάκη για το, για το, στον κύριο Κούς ε, για τρία λεπτά από το ID. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε και για την έκθεση. Δεν κατάφερα να διαβάσω την έκθεση, οπότε δεν θα εκφέρω γνώμη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κούς. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να πάρει τον λόγο για να ρωτήσει κάτι, να σχολιάσει από τους συναδέλφους. Αν όχι, να καλωσορίσω αμέσω το προσκεκλημένο μας, τον κύριο Μάριο Φάρκστερτ, τον οποίο ευχαριστώ για την παρουσία του εδώ στην Επιτροπή. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα σας δώσω αμέσως το λόγο και σας παρακαλώ να περιοριστείτε στα πέντε λεπτά. Στην κυρία, συγγνώμη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Αϊκάουτ και τους κοιοδησίτες που κατέθεσαν τις απόψεις τους επί του ελέγχου των δραστηριοτήτων της Τράπεζας του 2018. Χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι εδώ και έχω τη δυνατότητα να σχολιάσω μερικά από τα όσα είπατε. Χαίρομαι, διότι είμαστε η μόνη, ο μόνος πολυμερής ε, αναπτυξιακό οργανισμός ο οποίος ε, έχει τέτοιο διάλογο, δημοκρατικό διάλογο με ένα εκλεγμένο κοινοβούλιο. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο για μας, είναι εξαιρετικά χρήσιμο για άλλου του ε, μπλεκομένου μα του μετόχου, ΜΚΟ κλπ. Αυτό μα βοηθάει πράγματι πολύ. Επίσης, αποτελεί συνέχεια τη συνεργασία με άλλες επιτροπές τον περασμένο μήνα για παράδειγμα. Είχαμε εξαιρετικές συνομιλίες, συζητήσεις με τους αδέλφους σας από την ΕΚΟΝ και την BADGE. Έρχομαι σε αυτά που είπατε. Είπατε, περισσότερη δημοσιοποίηση στοιχείων σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση. Ναι, το κάνουμε. Ίσως όχι ε, με την απαιτούμενη διαφάνεια που θα θέλατε, αλλά υποβάλλουμε έκθεση, αυτό που λέει και ο εισηγητής και θα συνεχίσουμε φυσικά να το κάνουμε όλο και καλύτερα. Επίσης, ναι, είμαστε στο 2020 και συζητούμε ακόμη το 2018. Ε, έκτοτε συνέβησαν ένα σωρό καλά πράγματα, καλά για την ΕΤΕΠ και τους πολίτες μας. Είμαστε λοιπόν στο 2020, κατά τη διάρκεια του οποίου θα δούμε και άλλες καλές εξελίξεις. Ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στη Συμφωνία των Παρισίων. Θα σας πω τι σημαίνει αυτό για την πολιτική που εφαρμόζουμε. Επίσης ε, εργαζόμαστε για την πολιτική μεταφορών. Συνεχίζουμε το έργο μας στο θέμα των προτύπων περιβαλλοντικής κοινωνικής και γενικότερης διακυβέρνησης η πολιτική μας κατά της απάτης θα αναθεωρηθεί. Ε, θα συμβούν πολλά καλά πράγματα κατά τη διάρκεια του 2020 και είναι κρίμα που κατά κάποιο τρόπο που ακόμη σχολιάζουμε το 2018. Εν πάση περιπτώσει, αν δούμε λίγο την γεωγραφική κατανομή των δραστηριοτήτων μας, θα έλεγα το εξή, ε, γιατί είναι σημαντικό το θέμα. Φυσικά δημοσιεύουμε στοιχεία. Αν δείτε μόνο τα κλασικά δάνεια, η κατάσταση μπορεί να σας φανεί λίγο παράδοξη. Αν όμω συγκρίνετε με το ΑΕΠ της κάθε χώρα, θα δείτε ότι η εικόνα είναι εντελώ διαφορετική. Ας πούμε το 19, οι χώρε ψηλά στον κατάλογο, από πλευρά ΑΕΠ, είναι η Ελλάδα, η Κροατία, η Κύπρος, η Πολωνία, η Λετωνία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Μάλτα. Βλέπετε ότι πρέπει να συγκρίνει κανείς με το ΕΠ για να καταλάβει κανείς πού βρισκόμαστε και τι σημαίνει αυτό για τα δάνεια και τις δραστηριότητε μας στις χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, η ΕΤΕΠ να γίνει μια ισχυρότερη τράπεζα προς την κατεύθυνση του κλίματος, ναι. Όχι να γίνει μια τράπεζα για το κλίμα, να γίνει μια ισχυρότερη τράπεζα για το κλίμα. Αυτό θέλω να πω. Γιατί ήδη από το 19 δανείζουμε πολύ περισσότερα σε συνάφη με το κλίμα εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τεδενιακή πολιτική στον τομέα των μεταφορών, τα είπα νομίζω, θα αναθεωρηθεί αυτή η πολιτική φέτος. Παρακολουθούμε επίσης ε, πώς θα να συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακολουθούμε τη νέα προσέγγιση του του τομέα των μεταφορών που θα, καταστρωθεί αργότερα φέτο. Και για την εταιρική διακυβέρνηση τώρα. Πέρσι, μετά από την αύξηση κεφαλαίου της ΕΤΕΠ, έγιναν επίσης πολλά στον τομέα της εταιρική διακυβέρνηση και θα συνεχίσουμε να αναθεωρούμε τον κώδικα διαντολογίας, για το Διοικητικό Συμβούλιο, για την Επιτροπή Διαχείρισης και ούτω καθεξής. Όσον αφορά τα δύο φύλλα, θα σας πω ότι από 18% είμαστε στο 30% γυναικών στην ανώτατη διοίκηση μεταξύ των ανώτατων διοικητικών στελεχών. Πολύ σημαντική πρόοδος, αν το καλοσκεφτείτε, το γίνει μέσα σε δύο χρόνια. 54% ε, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι γυναίκες. Στην Επιτροπή Διαχείρισης πάλι έχουμε τρεις γυναίκες ε, επί συνόλου εννέα. Λοιπόν, βελτιωθήκαμε, ναι, δεν ε, πετύχαμε όλους τους στόχους μας. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ε, στο προσωπικό μας γενικότερα, αλλά έχουμε στρατηγική και την ε, υλοποιούμε με στιβαρό τρόπο για να βρούμε τους ταλεντούχους ανθρώπους που θέλουμε για να έχουμε μια ισχυρή διοικητική δομή. Δύο θέματα πολιτικής μένω να σχολιάσω. Το ένα, η ΕΛΕΜ θέματα απόδοσης και προσθετικότητας, αν θέλετε. Ξέρετε, σας αφουγκραζόμαστε. Μαζί με την Παγκόσμια Τράπεζα αναλύσαμε έργα στην Αφρική και δημοσίευσαμε φως έκθεση όπου αξιοποιήσαμε ερευνητές από τη χώρα για να υπάρχει μεγαλύτερος αντίκτυπος. Αυτά δημοσιεύονται στη σχετική έκθεση, αυτά τα μπορεί να διαβάσει ο καθένας. Επίσης είμαστε πολυδραστήριοι σε χώρες χαμηλού εισοδήματος. Και θέματα διακυβέρνησης, χρηματοπιστικής διακυβέρνησης, θέλουμε να αλλάξουμε και σε αυτό. Γιατί ο αριθμός των μικρών εταιριών, των μικρών έργων, μας βοήθησε να βελτιώσουμε το μηχανισμό χορήγησης δανείων. Και αυτό έγινε χάρη στην εγγύηση των τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει με τις δικές μας κεφαλαϊκές απαιτήσει. Ελπίζω να τα κάλυψα όλα, κυρία Πρόεδρε, αλλά αν υπάρχουν ερωτήσεις, εννοείται, είμαι εδώ για να απαντήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριο Φαλκστέντ, ζητώ συγγνώμη για το λάθος που έκανα προηγουμένως ε, για την παρέμβασή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις ή άλλε σκέψεις, σχόλια. Αλλιώς ε, προτείνω να δώσουμε αμέσω το λόγο στον εκπρόσωπο της στην εκπρόσωπο ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Μερέτε Κλάουζερ, που είναι τμήματάρχη σε συντονισμό με τον όμελο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων από την Γενική Διεθνή Σιτσφέν. Έχετε λοιπόν αμέσω το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή. Ήταν πολύ καλή και πλήρης η έκθεση που μας παρουσίασε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ ικανοποιημένη, θέτει πολλά ζητήματα, πολλά ερωτήματα για πολλά σημεία πάνω στο οποίο θα συνεργαστούμε στενά και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και άλλους ενδιαφερόμενους. Θα περιοριστώ σε απαντήσεις που θα δώσω σε ζητήματα που θίξατε σήμερα. Για παράδειγμα, ακούσαμε παρατηρήσεις από την κυρία Κρετού η οποία είπε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή είναι κάτι πολύ σημαντικό, να μην ξεχνάμε χώρες και περιφέρειες που έχουν μείνει κάπως πίσω και χρειάζονται την υποστήριξή μας. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Ξέρουμε ότι υπάρχει και μια σημαντική κοινωνική διάσταση στους στόχους της πράσινης ανάπτυξης. Οπότε τονίζω ότι αυτό το οποίο θα γεφυρώσει τις διαφορές και θα τις μειώσει είναι ακριβώς η δίκαια μετάβαση. Κάτι το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μαζί ετοιμάζουν η Επιτροπή πρότεινε το μηχανισμό Δίκαια μετάβαση με στοχευμένη στήριξη προκειμένου να υπάρξουν κατάλληλε επενδύσεις προς τις περιφέρειες και τις χώρες αυτές. Αυτό το πρόγραμμα ε, μετάβαση θα προσφέρει ε, χρήματα, κονδύλια και επιχορηγήσεις και από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα για παράδειγμα από το Invest EU, που θα επικεντρωθεί στους στόχους της δίκαιας ε, μετάβασης, προσπαθώντας να συμπληρώσει τις επιχορηγήσεις οι οποίες θα διατεθούν. Και υπάρχει και εταιρική σχέση με την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που θα επικεντρωθεί αυτή τόσο στο τμήμα Invest EU, όσο και στη μόχλευση ε, δημοσίων κονδυλίων πράγματα που αναφέρονται και στην έκθεση. Κατά τη γνώμη μας έτσι θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Επίσης θέλω να επιβεβαιώσω ότι πράγματι ότι η στρατηγική για τις μεταφορές μας αναθεωρείται τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε να είναι έτοιμη στα τέλη της χρονιάς. Θα γίνει και αξιολόγηση επίσης της Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές. Θα πάει στην αξιολόγηση τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αρχίσουμε ήδη να κοιτάμε την αναθεώρηση της πολιτικής μεταφορών της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Φέτος δηλαδή, με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στις μεταφορές, την ε, ΤΕΠ κλπ. θα καταφέρουμε περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κλάζαν. Δεν ξέρω αν ο εισηγητής, ο κύριος Έκχαουτ, θέλει να προσθέσει κάτι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και την Κομισιόν. Ευχαριστώ για την ωραία αυτή συζήτηση. Βλέπουμε τι αλλαγέ όντω ε, το λεφτό προς την ΕΤΕΠ. Ξέρουμε ότι τα πράγματα αλλάζουν ακόμα και τώρα που μιλάμε. Γι' αυτό και δεν περιοριζόμαστε μόνο στο 18. Πάντως, δύο πράγματα πρέπει ακόμη να συζητήσουμε το οποίο θα δούμε τους, τα οποία προέκυψαν τη συζήτηση με τους ασκιώδες. Δεν βλέπω και μεγάλες διαφορές μεταξύ των θέσεών μας. Όμως, η κυρία Κρέτσου, για παράδειγμα, είπε να μην ξεχνούμε τις παλιές προτεραιότητες όταν μιλάμε για νέες προτεραιότητες. Αυτό νομίζω, σε αυτό νομίζω και η Κομισιόν. Ε, δεν νομίζω ότι είναι αντιφατικά αυτά τα δύο για μένα πρέπει να συνδυαστούν, να συγκεραστούν, να προχωρήσουν παράλληλα. Και, και αυτό γίνεται ούτως ή άλλως, πιστεύω. Άρα, να μην δημιουργήσουμε μια τεχνητή αντίθεση μεταξύ παλαιών και νέων προτεραιοτήτων εκεί που δεν υπάρχει. Αν υπήρχε θα το έλεγα, αλλά δεν βλέπω κάποια αντίφαση εδώ. Γι' αυτό και λέω στην αρχή του κειμένου για την γεωγραφική ισορροπία, το είπε και η κυρία Γκινέα, να υπάρχει γεωγραφική ισορροπία. Αυτό το επικρίνω στην έκθεσή μου, γιατί αν δεν λάβει κανείς υπόψη του το ΑΕΠ θα καταλήξει μια τεχνητή εικόνα, σε μια ψευδή εικόνα. Νομίζω η ΕΤΕΠ το σχολίασε και απήντησε από αυτού, αναφέροντας δηλαδή τη, τη σχέση δανείων ως προς το ΑΕΠ της κάθε χώρας, που είναι και το σημαντικό. Πάντω, σε κάθε περίπτωση, η γεωγραφική ισορροπία είναι σημαντική. Να ξέρουμε λοιπόν ποιου βοηθούμε περισσότερο. Και για την δική μετάβαση, τη λεγόμενη δίκαιη μετάβαση, όπω είπε και η Επιτροπή, λίγο προσοχή εδώ, γιατί είναι όρος της μόδας. Όλοι μιλούν για δίκαιη μετάβαση, όμως δεν εννοούμε όλοι το ίδιο πράγμα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για έναν μηχανισμό δικής μετάβασης, μιλούμε για τις περιοχές που είναι σε μετάβαση και όπου οι άνθρωποι εντό τη συγκεκριμένη περιοχή εκτίθεται σε διαφορετικές επιπτώσει. Αλλά μπορεί να μιλούμε επίση για τη χρηματοδότηση. Άλλο θέμα. Ε, ποια είναι η μετάβαση που πρέπει να γίνει στη βιομηχανία. Καινούριο θέμα αυτό. Και το λέω προ το ΕΛΚ που λέει μην ξεχνάμε τη βιομηχανία. Ναι. Το μέλλον της βιομηχανίας μας είναι μια πράσινη βιομηχανία και εκεί πρέπει να επενδύσουμε βεβαίως. Και αυτό πρέπει να γίνει με δίκαιο τρόπο. Θέλω να πω ότι κάθε φορά που λέμε δίκαιη μετάβαση έχουμε πολλές διαφορετικές μεταβάσεις. Δεν είναι όλα η ίδια δίκαιη ε, μετάβαση και δεν είμαι καθόλου αντίθετος εννοείται. Αλλά προσοχή όταν χρησιμοποιούμε τον όρο δίκαιη μετάβαση. Άλλο το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, άλλο η ΕΤΕΠ και ούτω καθεξής. Διαφορετικές προσπάθειες. Για τις μικρομεσαίες, χαίρομαι, σημαντικό θέμα. Δεν κατάλαβα καλά αυτό που είπατε, περισσότερη διαφάνεια, είπατε που θα οδηγήσει σε γραφειοκρατία, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα ποιο είναι, ποιος είναι προβληματισμός. Και εδώ ίσως να μην έχουμε την αντίφαση που που περιγράψετε. Και η τελευταία ζήτηση που πρέπει να έχουμε είναι τι εννοούμε όταν λέμε ευθυγράμμιση, εναρμόνιση με το Παρίσι, με τη Συμφωνία των Παρισίων. Γιατί εκεί θα αρχίσουμε να μιλάμε για τα αερία για τις πολιτικές δανείων, για την πολιτική επενδύσεων, τα δικαιώματα κλπ. Ευθυγράμμιση με το Παρίσι σημαίνει ισοσκελισμένο ισοζύγιο, ουδέτερο ισοζύγιο για το 2050 να το συζητήσουμε αυτό, αλλά αν μιλάμε για το 2050, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ μιλάμε για επενδύσεις σήμερα, αύριο το πολύ. Δηλαδή, να επενδύσουμε σήμερα με γνώμονα και έχοντα στο μυαλό μα φυσικά το που πρέπει να βρισκόμαστε το 2050. Αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το λεφτό για να πω ότι δεν είναι σαφέ τι εννοούμε όταν λέμε ευθυγράμμιση με το Παρίσι. Ξέρουμε πότε μια δαπάνη συνάδει προ την προστασία του κλίματο, αλλά ευθυγραμμίσει με το Παρίσι είναι λίγο γενικό και αόριστο. Ούτως ή άλλως η αλλω η συζητηση δεν έχει καταλήξει, έτσι. Γι' αυτό λέω και αυτό να το συζητήσουμε ευρύτερα ω κοινωνία, έτσι ώστε στην συνέχεια να μπορέσουμε να συζητήσουμε και τι συγκεκριμένε πρωτοβουλίε στο πλαίσιο του Παρισιού. Αν θέλετε να αλλάξω τη διατύπωση, δεν έχω κανένα πρόβλημα. αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι ευθυγραμμισμένα με το Παρίσι. Δεν καταλαβαίνουμε όλοι το ίδιο ε, πράγμα τα λέμε ευθυγράμμιση με το Παρίσι. Και το τελευταίο τελευταίο, μια που έχουμε και την Κομισιόν εδώ, η έκθεσή μου προφανώς αφορά την ΕΤΕΠ και την ε, διαφάνεια και την διακυβέρνηση, αλλά μια που είμαστε εδώ όλοι, και συζητούμε και τις μελλοντικέ πολιτικές δανείων, νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο η Κομισιόν ορίζει τα διοικητικά στελέχη της ΕΤΕΠ. Γιατί καλή ενέργεια, ε, καλή και συζήτηση για τον τομέα των μεταφορών. Λοιπόν, ποιες θέσεις παίρνει η Κομισιόν στα διοικητικά όργανα της ΕΤΕΠ. Θα ήθελα και εδώ περισσότερη διαφάνεια. Διαφάνεια όσον αφορά τι θέσει, τη στάση που κρατάει η Κομισιόν στα διοικητικά όργανα τη ΕΤΕΠ. Αυτό αφορά την Κομισιόν, επαναλαμβάνω. Γιατί την συνεχεία η Κομισιόν λογοδοτεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δράτω με τη ευκαιρία <laughs> να το πω προφορικό τρόπο έχουμε τον Κομισιόν. Δεν μπορώ να το πω στην έκθεση γιατί αφορά την ΕΤΕΠ, αλλά πραγματικά θα θέλαμε ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δούμε μια βελτίωση εδώ. Διαφάνεια στην στάση που κρατάει η Κομισιόν στα διοικητικά όργανα τη ΕΤΕΠ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, μικρομεσαίε επιχειρήσει, ε, Παρίσι, γεωγραφική κατανομή, θα τα βρούμε όλα αυτά. Αυτά είναι τα βασικά θέματα σίγουρα θα συνεχίσουμε και θα βελτιώσουμε τον διάλογο στο μέλλον και πιστεύω ότι πραγματικά η ΕΤΕΠ θα γίνει μια πραγματική τράπεζα για το κλίμα, μια καλύτερη τράπεζα για το κλίμα. Έτσι το περιγράφω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Εικχάουτ για τη ε, σχόλιά σας και σας ευχαριστούμε κυρίως και για τη δουλειά που κάνατε και για τις προσπάθειες που θα καταβάλλετε ακόμη για αυτή την έκθεση. Ήθελα να επενθυμίσω ότι η προθεσμία υποβολή τροπολογιών για αυτή την έκθεση είναι η 3η Μαρτίου του 2020 στις 2 το μεσημέρι. Ευχαριστώ ξανά όλους τους συναδέλφους που παρευρέθησαν σήμερα στην Επιτροπή. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, την κυρία Φάλξτετ, την κυρία Κλάουζεν, εκ μέρους της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ για τα όσα μας είπατε, για τη δουλειά που έχει ήδη γίνει.